przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Beginning of the έναρξης της Συνόδου της Ολομελίας.